ομάδα ALDE, GUE, ELK, ECR και EFDD έλαβα ε, προτάσεις για αλλαγέ στις ε, θέσεις των, στις Δημοσιεύονται λοιπόν αυτό στα πρακτικά. Αν δεν θεωρηθεί, αν δεν υπάρξουν ενστάσεις, θεωρούνται οι αλλαγέ αυτές εγκεκριμένες. Και τώρα να σας πω ποιες είναι οι προθεσμίες για την υποβολή τροπολογιών για τον